Cari colleghi, diamo inizio alla... Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε το τμήμα της συνεδρίας μας που αφορά τις ψηφοφορίες. Πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, μπορώ να σας ανακοινώσω ότι η Οικονομική Επιτροπή διαβίβασε μια τροποποίηση στο κείμενο που διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα δημοσιευτεί η τροποποίηση, η διόρθωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 4 του εσωτερικού κανονισμού, η διόρθωση αυτή θεωρείται εγκεκριμένη εκτός εάν εντός 48 ώρου μια πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 βουλευτές δεν επιθυμούν να τεθεί σε ψηφοφορία. Είμαστε έτοιμοι για τις ψηφοφορίες. Απλουστευμένη διαδικασία για την έκθεση Ρέουλ σχετικά με την ε, ένταξη της ευρωπαϊκής κοινότητας ε, στην ε, υπηρεσία, στη διεθνή υπηρεσία για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται τώρα. Avete votato tutti? Ψηφίσατε όλοι. C'è una parte che dice sì e una parte dice no. Bisogna essere Κάποιοι λένε ναι, κάποιοι λένε όχι. Ε, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη έτσι. Adesso credo che abbiate votato tutti. Τώρα νομίζω ψηφίσατε όλοι. Bene, dichiaro chiusa la votazione. Πέρα τη ψηφοφορία. Votanti in totale 470. Εψήφισαν 478 υπέρ 453 ε, κατά 13 αποχές 12. Εγκρίνεται η έκθεση. Ζήτησε το λόγο ο κύριος Καζίνη παρακαλώ. Δεν πρόλαβα. Αν είχα προλάβει όμως θα υπερψήφιζα. Μάλιστα. Ωραία. Να προσμετρηθεί άλλη μία ψήφος λοιπόν. Αυτή του συναδέλφου Καζίνη. Λοιπόν, πάλι απλουστευμένη διαδικασία για την έκθεση Δεκάστρο. Κατάργηση κάποιων αποχαιωμένων κανόνων του Συμβουλίου στον τομέα της ε, κοινής ε, γεωργικής πολιτικής. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται τώρα. Avete votato tutti? Ψηφίσατε όλοι. Καλώς πέρας της ψηφοφορίας. Βοτάντι 543. Εψήφισαν 543. Υπέρ 542. Κατά μία ψήφος αποχή μη δεν. Συντριπτική πλειοψηφία. Βουλγαρική όπως τη λέμε εμείς. Βουλγαρική. Αλλά όχι στη σημερινή Βουλγαρία που είναι απόλυτα δημοκρατική χώρα, Της παλαιάς. Ψηφοφορία σύμφωνα με απλουστευμένη διαδικασία για την έκθεση Ντεκάστρο για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων για τι εργαστηριακές αναλύσεις. Ονομαστική ψηφοφορία. Avete votato tutti? Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εψήφισαν 577. Υπέρ 534. Κατά 29. Αποχές 14. Εγκρίνεται η έκθεση. Relazione dell'onorevole Hubner, sempre secondo la procedura. Έκθεση Hübner Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται τώρα. Εψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. Εψήφισαν 604 υπέρ 579 κατά 13 αποχές 12. Εγκρίνεται. Ο Στάφος Μάρτιν θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, θα ήθελα να πω ότι και εμένα δεν λειτουργήσε η δική μου συσκευή και εγώ ήθελα να ψηφίσω ναι, να υπερψηφίσω. Σημειώνουμε. Κύριε Μαρτίν, τα λεγόμενά σας. Πάμε στο επόμενο, πάντα προσθεμένη διαδικασία, Γκέριγκερ, για τα άγρια πουλιά. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Votanti 619, favorevoli 590. Ψήφισαν 619, υπέρ 592, κατά 4, απόχέ 23. Εγκρίνεται η έκθεση Γκέρινγκ. Δεύτερη έκθεση Γκέρινγκ. Πάντα με απλωστευμένη διαδικασία. Ε, εξοπλισμοί που λειτουργούν με φυσικό αέριο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 638, 618. Ψήφισαν 638 υπέρ 618 κατά 11 αποχές 9. Εγκρίνεται η έκθεση Γκέριγκερ. Τρίτη έκθεση Γκέριγκερ για την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Άρχεται η ψηφοφορία. Avete votato tutti? La votazione è chiusa. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εψήφισαν 641 υπέρ 620 κατά 13 αποχές 8 εγκρίνεται η έκθεση. Τέταρτη έκθεση Γκέριγκερ. Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας. Απλουστευμένη διαδικασία. Άρχεται η ψηφοφορία. Avete votato tutti, la votazione è chiusa. Πέρα τη ψηφοφορία. Votanti 654 favorevoli 643. Ψήφισαν 654 υπέρ 643, αποχές 11, ψήφι κατά 0. Συγχαρητήρια κυρία Γκέριγκερ για, για τέταρτη φορά. Πέμπτη έκθεση Γκέριγκερ, πάντα πλουστευμένη διαδικασία. Κτηνιατρική έλεγχη των ζώων που προέρχονται από τρίτες χώρες. που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Εψήφισαν 657 υπέρ 644 σαν κατά 11 δύο αποχές. Εγκρίνεται. Έκτη έκθεση Γκέριγκερ. Δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης επί των νοσοδημάτων και της οικονομικής λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων απλουστευμένη πάντα διαδικασία και ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινά τώρα που ολοκληρώνεται τώρα εψήφισαν 657 υπέρ 632 κατά 17 αποχές 8 εγκρίνεται 7η έκθεση Γκέριγκερ όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τι ενδοκινητέ συναλλαγέ και τι αγωγέ πουλερικών και αυγών για επόαση. Από τρίτε χώρε ε, θέτω σε ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία, την έκθεση. Πέραση Πέρασε ψηφοφορία. Ψήφισαν 662 υπέρ 641 κατά 15 Έξι αποχές. Εγκρίνεται και αυτή η εκθεση όγδοη 8η έκθεση Γκέριγκερ σχετικά με τα καθαρόαιμα βοηδή αναπαραγωγής. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. ψηφοφορίες. Ψήφισαν 655 υπέρ 633 κατά 13 9 αποχές. η συνάδελφος Γκέριγκερ έφερε σε αίσιο πέρας εννέα εκθέσεις. Σχεδόν ρεκόρ. Παρακαλώ, χειροκροτήσατε. Περνάμε τώρα στον κύριο Μπουσούτιλ, Σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυρικίου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχία διανομή. Απλουστευμένη διαδικασία, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Ψήφισαν 662 υπέρ 602 κατά 32 28 αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερη έκθεση Μπουσουτήλ για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϊχελών για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση για βραχία διαμονή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Ψήφισαν 667, υπέρ 610, κατά 28, αποχές 29. Εγκρίνεται η έκθεση. Τρίτη έκθεση Μπουσουτήλ συμφωνία απαλλαγή για την υποχρέωση θεώρηση για βραχία διαμονή μεταξύ κοινότητα και Μπαρμπάντο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Ψήφισαν 663 υπέρ 604 κατά 29 αποχές 30. Εγκρίνεται και η τρίτη έκθεση Μπουσουτήλ. Πάμε στην τέταρτη έκθεση Μπουσουτήλ. Πάλι απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση για βραχία διαμονή μεταξύ κοινότητα και Αγίου Χριστόφορου και Νέβη. Άρχεται η ψηφοφορία. La Πέρα τη ψηφοφορία. Ψήφισαν 664 υπέρ 603 κατά 28, 33 αποχέ. Εγκρίνεται η έκθεση. Σουτήλ e Πέμπτη έκθεση Μπουσουτήλ. Συμφωνία για απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ κοινότητας και Αντίγουα και Μπαρμπούντα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, Μπαρμπούντα, ε, όχι Μπάρμπα, δηλαδή η γενιάδα του κυρίου Σούλτς, έτσι. Πέρα τη ψηφοφορία. Ψήφισαν 672, υπέρ 612, κατά 29, αποχέ 31. Εγκρίνεται. Έκτη έκθεση Μπουσούτιλ σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση για βραχία διαμονή μετα... και την αντίστοιχη συμφωνία μεταξύ της κοινότητα και α, την Βρετανική Κοινοπολιτεία. τη Μπαχάμες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Ψήφισαν 672 υπέρ 608 κατά 31 αποχές 33 εγκρίνεται και αυτή. Συγχαρητήρια κύριε Μπουσουτήλ. Για την έγκριση, για την υιοθέτηση έξι εκθέσεών σας στην συνεδρία αυτή της Ολομελίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάμε τώρα στην έκθεση Χάουγκ διορθωτικός προπολογισμός υπαρθμών 9 του 2009 για τον σεισμό στην Ιταλία. Άρχεται η ψηφοφορία, χρειάζεται ειδική πλειοψηφία. Πέρας της ψηφοφορίας. Ψήφισαν 673 υπέρ 654 κατά 4 αποχές 15 εγκρίνεται η έκθεση Χάουγκ. Ευχαριστώ κυρία Χάουγκ και στο όνομα της Ιταλίας το λέγω αυτό. Πάμε τώρα στην έκθεση Μπόγκε για την κοινοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή και Παγκοσμιοποίηση ονομαστική ψηφοφορία χρειάζεται ειδική πλειοψηφία. Άρχεται η ψηφοφορία. La votazione chiusa. Πέρας της ψηφοφορίας ψήφισαν 677 υπέρ 598 κατά 49 30 αποχές. Συγχαρητήρια, κύριε Μπόγκα. Προβάτα. Πάμε στην έκθεση Wallis. Έτηση άρσης της ασυλίας του Μάρεκ Σίβιετσα. Άρχεται η ψηφοφορία. E chiusa τη ψηφοφορία ψήφισαν 671 υπέρ 639 κατά 17, 15 αποχές. Εγκρίνεται η έκθεση. Έκθεση Κοέλιο. Μηχανισμός αξιολόγησης για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σέγγεν. Δεν υπάρχουν τροπολογίες. Την θέτω λοιπόν την έκθεση ως έχει σε ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Stiamo votando la proposta di decisione sulla quale Ψηφίζουμε για την πρόταση επί της οποίας δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Όχι.